καθυστέρηση. Εφόσον ε, είναι παρόν ο εισηγητής θα μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έκθεση David Martin για την προσαρμογή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Κύριε David Martin, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, ανεκτικότητα και την παρουσία σας. Όταν το 1984 έγινε για πρώτη φορά μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπα στους συνοδέλφους τότε και ειδικότερα στον Κέτ Γόεν, Σκοτσέζο συνάδελφο ότι δεν ήξερα μήπως είχα κάνει λάθος επιλογή διότι φαίνεται να έχει και πολλή αρμοδιότητα σε νομοθετικά θέματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τώρα όμως, όταν ρωτήσει κανείς τη μητέρα ο οποιοδήποτε νεαρού παιδιού, ε, εκείνη θα σας πει ότι το παιδί μπορεί να, να, εντυπωσιάσει μόνο, έστω, παρόλο που δεν έχει δόντια, ε, πολύ καλά και με τα ούλα του. Κάτι λοιπόν το ίδιο πιστεύω ότι συνέβη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συνθήκη της Λισαβόνας θα επιτρέψει πλέον στο Κοινοβούλιο να ενηλικιωθεί πλήρως, να αποκτήσει και να χρησιμοποιεί όλα τα δόντια του και να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σαν οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο. Χαιρετίζω τις νέες εξουσίες που θα αναλάβουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά θέλω να πω ότι είμαι και λίγο απογοητευμένος διότι αυτή η έκθεση έπρεπε να ονομάζονταν η έκθεση Κόρμπετ. Ο συνάδελφος Κόρμπετ είχε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά πριν τις εκλογές πάνω σε αυτή την έκθεση. Δεν συμφωνούσαμε για, τα, για κάποιες όψεις που δεν είχαν σχέση με τη Λισαβόνα, αλλά για το θέμα της Λισαβόνας έκανε θαυμάσια δουλειά ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ και είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω αυτό θα υπάρξουν. Τώρα η έκθεση εστιάζεται στι εμπορικέ πολιτικές, θα έχουμε νέες εξουσίες στον τομέα τη και της Γεωργία, όπου θα υπάρχει πλέον συναπόφαση για το διορισμό των μελών τη ευρωπαϊκή Επιτροπή. δημιουργεί μια νέα σχέση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και Επίσης ε, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας σας πω τώρα που διαφωνούμε μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Οι πολιτικές ομάδες επέδειξαν θαυμάσιο πνεύμα συνεργασίας. Όλοι οι σκιώδεις ε, και συντονιστές ε, και, οι άλλοι, και, όλοι οι οι συγητές και οι, και οι συντονιστές και όλα τα μέλη των ομάδων ε, επαναλαμβάνω επέδειξαν θαυμάσιο πνεύμα συνεργασίας όταν συζητούσαμε θέμα όπως ε, του, Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ε, κάποιος, δεν συμφώνησαν όλοι, είπαν ότι ο αντιπρόεδρος θα πρέπει να είναι ο πρόεδρος της ΚΟΖΑΚ της οποίας πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες και σε ό,τι αφορά τη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια είχαμε κάποιες διαφωνίες για το βαθμό λεπτομέρειας στον οποίο θα έπρεπε να προχωρήσουμε πόσο πολύ πρέπει να διαγράφουν και να ορίζουν αυτή τη σχέση οι διατάξεις του κανονισμού. Ο κύριος Μπρόκ επέδειξε τη δέουσα ευελιξία για το θέμα αυτό ώστε να υπάρχει περιθώριο για εσάς να με τους ομολόγους των Εθνικών Κοινοβουλίων τις λεπτομέρειες της συνεργασίας μας με τα Ευρω... Εθνικά Κοινοβούλια, κύριε Πρόεδρε. Υπήρξαν και κάποιες διαμάχες για το θέμα της επικουρικότητας. Ο ρόλος των επιτροπών καθορίστηκε σαφώς. Δεν υπήρξε διαφωνία από αυτού. Το μόνο πρόβλημα ήταν τι θα συμβεί αν μια επιτροπή πει όχι παρεμβαίνει η επικουρικότητα και πρέπει να συνεχίσουμε το νομοθετικό μας έργο. Μήπως πρέπει να υπάρχει κάποια ασφαλιστική δικλίδα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ κατέθεσα τροπολογίες, ε, κατέθεσαν τροπολογίες και άλλοι. Ένα δέκατο των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρεί ότι υπάρχει θέμα επικουρικό, προκύψει θέμα επικουρικότητας. Αυτό πρέπει να συζητηθεί από την Ολομέλεια και εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια ικανοποιητική ασφαλιστική δικλίδα. Τέλος θέλω να αναφερθώ και στο θέμα των παρατηρητών πρέπει να έχουμε παρατηρητές. Εγώ λέω ναι, το σημαντικό θέμα και η Επιτροπή συμφώνησε από αυτού. Το σημαντικό θέμα είναι οι παρατηρητές, θα είναι οι άνθρωποι που αλλιώς θα κλαίγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό εδώ παίζεται η αξιοπιστία μας. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε δυνατότητα να επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε να αναλάβει θέμα παρατηρητών. Ορισμένοι πρότειναν τον διορισμό εθνικών βουλευτών. Εγώ δεν συμφωνώ επ' αυτού και θα ολοκληρώσω λέγοντας κύριε Πρόεδρε ότι από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουμε ένα σώμα κανόνων που θα μας επιτρέπει να ασκήσουμε άμεσα τις νέες μας εξουσίες. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας και θέλω ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω όλους μας, ε, μας βοήθησαν ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε πλέον αυτό το νέο κανονισμό Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή σας. Ευχαριστώ διότι μας παρουσιάσατε τη γνωμοδότησή σας σε σχέση με την έκθεση αυτή και τώρα εξ του ΕΛΚ ο κύριος Τάνκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές, βεβαίως ε, είμαστε ευτυχείς ε, που πρόκειται να ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, πήρε αρκετό χρόνο και δεν φταίει γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι άργησε να κυρωθεί. Άρα η άμεση δυνατότητα εφαρμογής δεν πρέπει να καθυστερήσει λόγω υπετιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τη στιγμή που θα είναι δυνατόν να μπορέσουμε να εξασκήσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα. Κατά αυτόν τον τρόπο το Κοινοβούλιο θα ενισχυθεί. Η συνθήκη της Λισαβόνας βελτιώνει σημαντικά τις δυνατότητες και ενισχύει τις δυνάμεις και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μπορέσει να προχωρήσει και να μπορέσουμε να να εξασκήσουμε όλα τα δικαιώματα που έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω ε, και τον κύριο Μάρτιν και τον κύριο Κόρβετ για την προσπάθειά τους ε, για ε, τα θέματα τα οποία εξήτασαν τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη ή τους πολύ αυστηρούς ελέγχους ή το ότι έχουν τονίσει περισσότερο την επικουρικότητα, τη δυνατότητα επιτροπολογίας και συναπόφασης και θα είμαι πολύ ευτυχής να, βλέ... να δω να υλοποιούνται όλες αυτές οι δυνατότητες αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν ε, θα καταχραστούμε τα δικαιώματα αυτά. Δεν πρέπει να είμαστε μία ε, μειονότητα η οποία θα καταχραστεί τα δικαιώματα αυτά για να επιβραδύνει την ε, νομοθεσία. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει ένας μοναδικός πρόεδρος να ε, οδηγήσει στην κατάρρευση το σύστημα. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λειτουργήσει για να μπορέσει να προχωρήσει και θέλω να συνεργαστώ τους συντάκτες της εκθέσεως. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Ραμόν Χαραγκουή Ατόντο έχει το λόγο. Εξ των Σοσιαλιστών και Ευρωπαίων Δημοκρατών και εγώ θα ήθελα να πω ότι για τη Σοσιαλιστική Ομάδα είναι μεγάλη τιμή το γεγονός ότι η Κόρπετ και Μάρτιν ήταν οι πρωταγωνιστές αυτού του εγχειρήματος και ελπίζω να γίνει αποδεκτό από ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μία πράξη ύψης της σημασίας και μεγάλες, μεγάλες εμβέλειες, διότι από την πρώτη δωδεκάτου θα ισχύσει και ο κανονισμός πέρα από τη συνθήκη. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσαρμοστεί για να έχει ένα μέσον αντιμετώπισης και ανταπόκρισης στη νέα συνθήκη. Νομίζω ότι συνοψίζοντας θα πρέπει να πούμε ότι η έκθεση μας βρίσκει σύμφωνος. Αλλά σε σχέση με τις εκρεμείς μεταρρυθμίσεις θα ήθελα να τονίσω τα εξής. Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση για το ποιες τροπολογίες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και ποιες όχι. Επειδή στρίκτο σένσου μιλάμε για μια συνθήκη, τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα ήθελα ο ίδιος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίσει κατά πόσο ορισμένες από τις, ε, ένα μέρος της αναθεώρησης του κανονισμού αρμόζει ή όχι. Δηλαδή, ο, αν το ορίσει ο πρόεδρος, εμεί θα το δεχτούμε. Όταν μιλάμε για αναθεώρηση ενός κανονισμού, θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία για ένα θέμα τέτοιας εμβέλειας. Άρα πριν από την Πέμπτη θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί των ε, τροπολογιών που θα ψηφίσει το Σώμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας ε, πω το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μετά από τις παρεμβάσεις των πολιτικών ομάδων, θα σας πω ποιες είναι οι διατάξεις που ε, διέπουν την ψηφοφορία αυτής της ε, έκθεσης όπως ορίζει η διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Άντριου Νταφ έχει το λόγο εξ ονόματος των ε, φιλελευθέρων. Άντριου Νταφ. Πρόεδρε. Η ομάδα ALDE χαίρεται που μπορεί να δεχτεί την έκθεση Corbett Martin. που θέτει το κοινοβούλιο σε ένα νέο δρόμο, σε μια νέα δίωδο, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προετοιμαστεί έτσι ώστε να αποτελέσει ε, μία πραγματική συνέλευση. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια τάχιστα και αποδοτικά για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα του ευρύτερου πολιτικού φάσματος. Ως προς την ε, αντιμετώπιση των εθνικών κοινοβουλίων, η συνθήκη πολύ σωστά προτείνει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας μεταξύ του Ευρωπαϊκού δηλαδή Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όμως η συνθήκη σιωπά είναι πολύ διακριτική ως προς τη συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε και να έρθουμε σε διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια για να δούμε ποια είναι η δική τους προσέγγιση του ζητήματος. Πώς ερμηνεύουν δηλαδή τη συνθήκη τα εθνικά κοινοβούλια πριν θέσουμε επιτάπητος λεπτομεριακά σχέδια. από μόνοι μας με βάση τις δικές μας διαδικασίες. Από την πείρα μας, υπό την αιγίδα της Κόζακ, η πείρα μας δείχνει μεγάλη διαφορά, μεγάλες διαφορές ως προς τις προσεγγίσεις των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας, με το ζήτημα της επικουρικότητας. Νομίζω λοιπόν Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά αυτή την, αυτές τις διαφορές και δεν θα πρέπει να επισημοποιήσουμε τη μεθοδολογία συνεργασίας. σε σχέση με την ε, χρήση του μηχανισμού επικουρικότητας στην παρούσα φάση. Πέραν αυτού, η ομάδα των φιλελευθέρων υποστηρίζει πλήρως τις ε, προτάσεις προτάσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταφ. Και τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων, το λόγο έχει ο κύριος Χάφνερ. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό το κοινοβούλιο είναι γρήγορο. Κάνει τα μαθήματά του, ε, δρά και πρέπει να πούμε ότι ε, χρειάστηκαν 7 χρόνια μέχρι ότου να ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνας αλλά για μας ε, επειδή το Κοινοβούλιο έχει ήδη προετοιμαστεί καλά μέσα σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε διεκπαιρεώσει τις υποχρεώσεις μας κατά τρόπον ώστε να έχουμε ενισχύει τον καινούριο εσωτερικό κανονισμό μόλις ισχύσει η συνθήκη. Θα πρέπει ε, να ε, περιοριστούμε εις ε, τα θέματα της αρμοδιότητός μας διότι πιστεύω ότι για τα υπόλοιπα θέματα θα έχουμε επαρκή χρόνο εδώ για να τα συζητήσουμε αλλά αυτό που είναι απαραίτητο πρέπει να διεκπεραιωθεί αμέσως και αυτές οι ε, ε, οι ρυθμίσεις θα επιτρέψουν να υπάρχει μία απλοποιημένη διαδικασία σύνομη με τη συνθήκη και φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια πράγμα το οποίο στηρίζουμε σε ορισμένα άλλα θέματα θα θέλαμε να προχωρήσουμε και περισσότερο παραδείγματο χάρη όσον αφορά την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κρόσα αλλά προς το παρόν θέλω να χαιρετήσω τι συμφωνίε και να ευχαριστήσω όλους τους ε, συνεισηγητέ. Ευχαριστώ. Και τώρα για δύο λεπτά θα δώσω το λόγο στον Ashley Fox τον εκπρόσωπο των, της ομάδας των Ευρωπαίων Μεταρρυθμιστών και Συντηρητικών. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διατυπώσω τις δικές μου ανησυχίες για το γεγονός ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε την τροπολογία Μπροκ για το καθεστώς των μελών. Ο Έλμε Μπρόκ είχε προτείνει τη μεταβίβαση ευθύνη από το Προεδρείο που θα συνεδριάζει μη δημοσίω στο Κοινοβούλιο που συνεδριάζει δημοσίω. Εγώ πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι μας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν όχι μόνο τι αμοιβέ εισπράττουμε, αλλά και τις λεπτομέρειες ε, των επιδομάτων και των άλλων ε, παροχών που έχουν Και λυπάμαι που εσείς σκέφτεστε, ω πρόεδρός μας σκέφτεστε διαφορετικά. Πιο ανησυχητικό ακόμα είναι η αγωνία να χάσουμε μία ψήφο ή και προκειμένου να γίνει ε, κάποια ψηφοφορία ακολουθείται διαδικασίες που κατά την άποψή μου δεν είναι δημοκρατικές. Μια εποχή που όλοι μιλάμε για το πώς θα γίνει πιο διαφανής η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πλησιάσει περισσότερο τους πολίτες της, η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από τεράστια υποκρισία. Αν θέλει να αυξήσει την διαφάνειά της η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργήσουμε να ενεργήσουμε δυναμικά και όχι να λέμε απλώς λόγια κενά περιεχομένου για αυτό το θέμα. Το να μην ε, ε, ε, δεν πρέπει να φερόμαστε στους συμπολίτες μας σαν μανιτάρια τα οποία θα τα σκεπάζουμε με με, με χώμα για να ζουν στο σκοτάδι και δεν θα τους επιτρέπουμε να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει εδώ που συνεδριάζουμε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Όλα μπορούν να συζητηθούν αγαπητέ συνάδελφε. Τίποτε δεν παραμένει κρυφό και σκοτεινό. Τίποτε, τίποτε δεν παραμένει κρυφό. Πρέπει όμως να πάρουμε τις αποφάσεις ε, τη μία μετά την άλλη τηρώντας τους κανόνες μας και τίποτε άλλο. Βεβαίως μπορεί όμως να υπάρξει για όλα τα θέματα συζήτηση. Γιατί η ψηφοφορία για την τροπολογία Μπρόκ επετράπησε στην Επιτροπή και έγινε δεκτή και όμως θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί να συζητηθεί στην Ολομέλεια αν θέλετε να το συζητήσετε, θα το συζητήσουμε μαζί μόλις ολοκληρωθεί η συνεδρίασή μας. Αλλά πρέπει τώρα να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που προβλέπεται για την Ολομέλεια. Ο Hans Πιτ Μάτιν, επόμενος ομιλητής, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Η δημοκρατία είναι το αντίθετο της επανάστασης και το λέω, και το λέω τώρα και απευθύνουμε σε εσά κύριε Πρόεδρε. Τι κάνετε εδώ, διαμορφώνετε ε, την ζωή των ανθρώπων οι οποίοι είναι δημοκρατικοί αλλά για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να δημιουργήσουν μία, ε, μία πολιτική ομάδα και τους απομονώνετε Αναφέρομαι στο άρθρο 102 με το οποίο επέτρεψε ε, να έχουν οι πολιτικές ομάδες έναν ε, συντονιστή. Προηγουμένως το ίδιο ισχύει για τους μη εντεταγμένους πράγμα το οποίο τώρα δεν ισχύει πλέον σας ε, έχω ε, στείλει μία επιστολή, μου απαντήσατε στα γρήγορα, αλλά θα ήθελα να την ξαναδιαβάσετε, διότι ένα κοινοβούλιο το οποίο ουσιαστικό ε, υποστηρίζω δεν μπορεί να γίνει ένα κοινοβούλιο Δευτέρα τάξεως, διότι σαν μη εντεταγμένοι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε εγκαίρως και να συμμετέχουμε ενεργά. Γι' αυτό θα έπρεπε να αλλάξει επίσης ο εσωτερικός κανονισμός και ο κύριος Κόρμπετ ε, ε, γιατί εφόσον ήταν ριζοσπαστικός και εκλεγμένος σαν ριζοσπαστικός κάθεται εδώ σαν ε, το Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Όπως ξέρετε συζητάμε τα θέματα τα οποία αναφέρατε. Βρισκόμαστε ακριβώς μέσα στη συζήτηση, οπότε μην προεξοφλείτε τα συμπεράσματα. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε και ξέρετε ότι οι μη εντεταγμένοι δεν πρότειναν έναν ε, υποψήφιο, ε, το ξέρετε, αλλά θα λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τώρα να εξηγήσω ένα πολύ βασικό θέμα. Η διάσκεψη των προέδρων των πολιτικών ομάδων αποφάσισε ότι δεν θα ψηφίσουμε την Τετάρτη, σχετικά με την έκθεση του κυρίου Μάρτιν τα θέματα τα οποία δεν άπτονται της συνθήκη της Λισαβόνας διότι θα πρέπει να συζητηθούν περισσότερο και διεξοδικότερα. Θα γίνει η ψηφοφορία την Τετάρτη και θα ασχοληθούμε με τα θέματα που άπτονται της συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή είναι η απόφαση της διασκέψεως των Προέδρων των πολιτικών ομάδων και θα την εφαρμόσουμε. Αυτή λοιπόν είναι η πληροφορία την ε, οποία έπρεπε να σας μεταδώσω. Και τώρα ερχόμαστε στους επόμενους ε, ομιλητές. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως αντιλαμβάνομαι και στηρίζω την απόφασή σας, αλλά δεν θέλουμε ε, να υπάρξει ε, μία βαβούρα, αν μπορώ να το εξηγήσω έτσι, την Δευτέρα. Γι' αυτό θα ήθελα παρακαλώ να κυκλοφορήσουν αύριο σε όλους τους ευρωβουλευτές ποιες είναι οι τροπολογίες που δεν συνάδουν με τη συνθήκη της Λισαβόνας για να ξέρουμε γέρος περί τίνος πρόκειται και να μην έχουμε διαμάχες την Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή άλλωστε ήταν και η δική μου πρόθεση. Αυτό θα κάνω. θα ήθελα να συναντηθώ με τον πρόεδρο Κασίνη και άλλους συναδέλφους για να τους δείξω αυτόν τον κατάλογο και να τον δείξω και σε εσά προσωπικά αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα διότι δεν είσαστε παρόν. Αλλά πρόκειται για καθαρά τεχνικό θέμα. Κάποιο άλλο, ο κύριο Μέντε Βίγκο. Την ίδια ανησυχία θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ όπως και ο εισηγητής για να διεξαχθεί η ψηφοφορία την Τετάρτη θα πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιες είναι οι τροπολογίες που δεν γίνονται αποδεκτές. Γι' αυτό θα θέλαμε να τις έχουμε μέχρι αύριο το πρωί. Ναι. θα σας απαντήσω τώρα. Οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έπρεπε να ετοιμάσουν αυτόν τον κατάλογο που τον παρέδωσαν πριν από δύο ώρες. Είναι πολύ ε, πρόσφατος κατάλογος που μόλις ετοίμασαν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Θα σας τον παρουσιάσω δε τώρα αμέσω. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρλο Κασίνη. Πρόεδρε, θα σεβαστούμε τις αποφάσεις σας, αλλά τη στιγμή που υπάρχουν, επιφυλά... υπάρχουν επιφυλάξεις για ορισμένες τροπολογίες, ε, δεν σχετίζονται άμεσα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω όμως ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έχει γενικότερες αρμοδιότητες να υποβάλει προτάσεις ως προς την τροποποίηση του κανονισμού. Είτε προταθεί από μεμονωμένους ε, βουλευτές, είτε από ομάδα. Στα πλαίσια λοιπόν μίας ε, ευρύτερης αναθεώρησης του κανονισμού σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας για να γίνουν ορισμένες διορθώσεις δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί απαράδεκτο, αυτές οι τροπολογίες να θεωρηθούν μη αποδεκτές δηλαδή, διότι ορισμένες τροπολογίες μεταφέρουν στον κανονισμό το πνεύμα της ε, Λισαβόνας. Και πολύ συχνά αναφέρονται στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Μιλάμε για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι του Συμβουλίου. Εμείς βεβαίως θα σεβαστούμε τις αποφάσεις σας, αλλά έκανα σκόπιμο να υποβάλω αυτή την παρατήρηση. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, ο κύριος Σάντορ Ταμπάτζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση δείχνει σαφώς πως έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μια διαδικασία σημαντική μεταρρυθμίσεων που δεν θα μπορεί να καλυφθεί με μια μοναδική έκθεση. Ευχαριστώ τον, τον κύριο Μάρτιν και τον κύριο Κορμπέτ και όλους τους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που εκκρεμούν που θα πρέπει νομικά να προσδιοριστούν στο μέλλον. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Με χαρά βλέπω ότι το Κοινοβούλιο δήλωσε σαφώς ότι υποστηρίζει τα θεμελιώδη, το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά ε, έχουν ζητηθεί παρεκκλήσεις από αυτό το χάρτη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα που είναι ανοιχτά, τα οποία δημιουργούν κάποιες ανησυχίες, θέματα που θεωρούνται ότι δεν ανήκουν ακόμα στο κοινοτικό και εκτιμένο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν κυρίως σε ό,τι αφορά τα θεμελιώ... το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να προσδιορίσουμε επακριβώς ποια δικαιώματα θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση. και το θέμα της γλώσσας στη Σλοβακία δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λένε ορισμένοι ότι δεν ενδιαφέρει την Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, ε, έχω έρθει εδώ ως δημοκράτης ως κάποιον που έχει αναλάβει δημοκρατική εντολή. Μια εντολή παρόμοια με εκείνη που έχουν όλοι όσοι εξελέγησαν στο Κοινοβούλιο. Βρίσκομαι μπροστά σας επίσης σαν κάποια που έρχεται από μια χώρα με περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχει πολλά να τονίσει σε ό,τι αφορά εκείνου που προσπαθούν να καταλύσουν, να καταλύσουν τα δημοκρατικά δικαιώματα. Είχα έρθει λοιπόν με εμπιστοσύνη εδώ, αλλά ως πρώτη φορά νεοεκλογήσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνω ότι αποκλείομαι από τις συναντήσεις των συντονιστών, ότι δεν έχω φωνή στη διάσκεψη των Προέδρων και ότι τα θέματα αυτά αποτελούν ε, αντικείμενο συζητήσεων και πολύ χαίρομαι που ακούω ότι προσπαθείτε να λύσετε όλα αυτά τα θέματα αλλά σας καλώ κύριε Πρόεδρε τα θέματα αυτά να τα ολοκληρώσετε, να τα λύσετε το ταχύτερο δυνατό διότι είναι σημαντικό η δημοκρατική εντολή αυτού του Κοινοβουλίου να γίνει σεβαστή και σας καλώ να συναντήσετε τους ε, μη εντεταγμένους οι οποίοι και αυτοί είναι δημοκράτες και θέλουν να δώσουν συνέχεια σε αυτό το θέμα. Ε, Ο κύριος Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι Μάρτιν, ε, θέλω να συγχαρώ για τα θέματα που περιλαμβάνει η έκθεση για τους στόχους που επιτύχαμε. Πρέπει να σας πούμε ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γίνει ένα πλήρες και ισότιμο κοινοβούλιο και έφτασε ε, στην θέση την οποία προέβλεπαν αρχικά οι συνθήκες ε, και οι πολιτικές ομάδες και ε, το Προεδρείο και θεωρώ ότι είναι βασική απόφαση των, της διασκέψεως των Προέδρων και των Επιτροπών. Ο, θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό να μην συνεργάζονται με πλήρη συνυπευθυνότητα οι εθνικές επιτροπές με τις ευρωπαϊκές επιτροπές. Θεωρώ ότι ε, ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έρχονται οι πρόεδροι και όχι οι αντιπρόεδροι αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το Κοινοβούλιο και η Ολομέλεια δεν μπορεί να κρίνει εάν είναι σωστές ή λανθασμένες οι αποφάσεις των υπηρεσιών. Θα έπρεπε να αποφασίσει η Ολομέλεια και μόνο έτσι θα μπορέσουν να προστατευθούν οι βουλευτές διότι διαφορετικά δεν μπορώ να δεχθώ να ε, περιορίσουμε τις ε, αρμοδιότητες των Ευρωβουλευτών εδώ. Ευχαριστώ. Ο Ρομπέρτο για 1,5 λεπτό. Με την ε, έγκριση της έκθεσης Μάρτιν, στην ουσία ανταποκρινόμαστε σε μία αδύρυτη ανάγκη, δηλαδή να εγκρίνουμε μία έκθεση που θα αποτελέσει συνέχεια, ε, μάλλον θα αποτελέσει εμπροστοφυλακή της συνθήκης της Λισαβόνας. Μιλάμε για μια νομοθετική διαδικασία, μια δημοσιονομική διαδικασία και μια θεσμική εξισορρόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας μιλήσω λοιπόν για την αναθεώρηση των συνθήκων και για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων που φέρουν ε, συγκεκριμένη ευθύνη για την ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης ε, νομιμοποίησης και όχι ενός γραφειοκρατικού βραχνά. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν οι τροπολογίες αυτές που σχετίζονται άμεσα με την έκθεση και μετά θα μπορέσουμε να εξετάσουμε την αναθεώρηση του κανονισμού μας εις βάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία ε, αποτελούν αναπόσπαστο έργο της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων και αναφέρομαι στο θέμα της ε, τροπολογίας που αφορά τους παρατηρητές. Θα πρέπει οι παρατηρητές να είναι πρόσωπα που έχουν εκλεγεί ε, μέσα στα πλαίσια των Εθνικών Κοινοβουλίων του Ευρωπαϊκού. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τους συζητητές, ιδιαίτερα τον κύριο Μάρτιν και βεβαίως τον κύριο Κόρμπετ και να πω σε σχέση με τις τροπολογίες του κανονισμού ότι θα πρέπει να τονίσουμε ένα σημείο που αφορά τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απορρέει από αυτόν τον κανονισμό και τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία σχετίζεται άμεσα με τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις δύο μορφές νομιμότητας, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία. Αυτή που απορρέει από τους μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μηχανισμούς ελέγχου, νομοθετικούς μηχανισμούς και από την άλλη πλευρά την δημοκρατική συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών. Γι' αυτό συμφώνω απόλυτα με τις προτάσεις. Δεν συμφωνώ με τον Σνάφο Ντάφο, ο οποίος λέει ότι πρέπει να αφήσουμε για αργότερα τους μηχανισμούς συσχετισμού με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει να υπάρχουν, πιστεύω, παράλληλα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και δέχομαι τις προτάσεις ιδιαίτερα του κυρίου Μπρόκ ως προς την εκπροσώπηση της ΚΟΖΑΚ και συμφωνώ με τις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Μπρόκ και άλλων συναδέλφων σε σχέση με την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με άλλες συναφείς υπηρεσίες. Μάριο Μάουρο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Μιλάμε για αλλαγή φύσης και εργασίας των θεσμικών μας οργάνων. Μιλάμε για νομοθετικούς μηχανισμούς που θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ευκαιρίες που μας προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πώς θα κινηθεί η κοινοτική μηχανή στο εγγύς μέλλον. Γι' αυτό, αυτό που είναι το πραγματικό διακύβευμα είναι η ενίσχυση του ομοσπονδιακού χαρακτήρα καθώς και του επικουρικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι καθοριστική σημασίας για το μέλλον μας, διότι δεν λάβαμε επαρκώς υπόψη σε αυτή τη φάση τη... τον πολίτη, τον πολίτη υπό την τελεολογική έννοια, διότι η διαδικασία στην οποία φτάσαμε είναι ικανοποιητική, η Ευρώπη πια μετράει για τη ζωή των πολιτών, αλλά αντί να βάλουμε τον πολίτη στο επίκεντρο της πολιτικής, δυστυχώς έχουμε χειραγωγήσει την επικουρικότητα για να προωθήσουμε τα θεσμικά όργανα και τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό η αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, είναι αποφασιστική σημασία. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα εποπτείας για να έχουμε μια πραγματική αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων που εξετάζει το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα σε σχέση με την τήρηση αυτής της αρχής της επικουρικότητας, που θα πρέπει να είναι σημείο εκκίνηση των θεσμικών οργάνων και όχι να ορίζουν τη ζωή των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ. Μέντες Δεβίγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για το παραδεκτό των ε, τροπολογιών, και το κατά πόσο μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Εσείς ε, αναφερθήκατε στον κύριο Καζίνη, δηλαδή σε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων. Εμείς είμαστε ένα κυρίαρχο όργανο και μπορούμε να αποφασίσουμε κατά πόσο μια τροπολογία είναι αναγκαία ή όχι. Βρισκόμαστε σε ένα νέο στάδιο εργασιών. Γι' αυτό θα ήθελα να, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εξουσίες, ε, με σύνεση βεβαίως, και να κάνετε αυτό που αναμένουμε όλοι από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα παρακαλέσω τον εισηγητή να πάρει το λόγο. Κύριε Ντέιβιτ Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στη συζήτηση και θέλω να επανέλθω αυτό που μόλις μας είπε ο κύριος Μέντες Ντεβίγκο. Ο κύριος Κασίνη πολύ σοφά είπε ότι υπάρχουν τροπολογίες που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Απολύτως καμία σχέση και θα, θα μπορούσα να δεχθώ ορισμένες να ψηφιστούν, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε μια χωριστή συζήτηση για το θέμα αυτό προτού περάσουμε στην ψηφοφορία. Θέλω να καταστήσω ωστόσο σαφές. Τίποτα να εμποδίζει τα μέλη να υποβάλουν ε, θέματα όπως αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Φόξ, αφαίρεση από το Προεδρείο κάποιων εξουσιών υπέρ των κρατών μελών. Δεν έχω καμία αντίρρηση να υποβληθούν σε συζήτηση όλα αυτά τα θέματα στο μέλλον. Αλλά στροπολογίες όπως ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τη συνθήκη της Αβώνας, αλλά έχει σχέση, όπως είπε ο κύριος Κασίνη, με το πνεύμα της εφαρμογής της συνθήκης της Αβώνας, διότι αλλάζει η σχέση με τις τα εθνικά κοινοβούλια ε, μετά από την ε, έναρξη ισχύω της ε, συνθήκης της Λισαβόνας το θέμα των αντιπροεδριών στις επιτροπές και τα θέματα που έχουν σχέση με τον Προεδρείο δεν είναι θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη συνθήκη της Αβώνας και γι' αυτό δεν πρέπει να μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα σταματήσει η συζήτησή μας και θα κηρύξουμε τη λήξη της απόψινής μας συνεδρίασης. Η ψηφοφορία για την έκθεση Μάρτιν θα γίνει την Τετάρτη και η επόμενη Σύνοδος Ολομέλειας θα συνέλθει από το πρωί από τις 9 μέχρι τη 1 και από τις 3 μέχρι ε, τα μεσάνυχτα. Έχετε την ημερήσια διάταξη στα έγγραφα της Συνόδου και στην ιστοσελίδα. Λύεται η συνεδρία.